ολοκληρώθηκε στην παρούσα φάση. Πρωτού περνάμε στο επόμενο θέμα τη σήμερα. Συντάξτε να κάνω μια ανακοίνωση. Όπω θα θυμάστε, ο πρόεδρο τη 14 Μαρτίου του 2017 αποφάσισε να εφαρμόσει, να επιβληθεί μάλλον κύριο κατά του Κοβριμί και κατά, λόγω α, α, σχολείων απαράδεκτων κατά των γυναικών. Τρία μέτρα περιλαμβάνει λοιπόν αυτέ οι κυριώσει. Καταρχά, απώλεια αποζημίωση, ημερήσει αποζημίωση για 30 ημέρε. Κατά δεύτερον, πέρα από το δικαίωμα ψηφοφορία στην Ολομέλεια αναστολή των κοινοβουλευτικών καθηκόντων για 10 ημέρες ε, στο Κοινοβούλιο ή σε επιτροπές ή σε αντιπροσωπείες του Κοινοβουλίου και τρίτον απαγόρευση για ένα έτος της εκπροσώπησης του Κοινοβουλίου για, σε διακοινοβουλευτικό επίπεδο ή σε επίπεδο επιτροπών ε, κατέθεσε ε, καταγγελία κατά της απόφασης αυτής ο κύριος Κορμεν Μίκε στις 27 Μαρτίου και χθε το Προεδρείο επιβεβαίωσε την κύριοση του Προέδρου. Και έτσι λοιπόν ξεκινάει η περίοδο των κυρώσεων. Περνάμε στο επόμενο θέμα τη τη διάταξη, την έκθεση για την έγκριση και υποπτία τη αγορά των μηχανοκίνητων οχημάτων και των μολυκουμένων του και των συστημάτων κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που θεωρίζονται για τα αρχήματα αυτά. Και καταρχάς θα δώσω το λόγο για τέσσερα, λόγο, τέσσερα λεπτά το λόγο στον κύριο